Ε, στη ε, επιστημονικά πειράματα. Η τρίμηνη προθεσμία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αρχίσει από αύριο 18 Ιουνίου. Τα συνοπτικά πρακτικά της παρούς συνεδρίασης θα διανεμηθούν στην επόμενη συνεδρίαση, στην επόμενη σύνοδο του Κοινοβουλίου και αν δεν διαφωνείτε τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στην παρούσα σύνοδο θα διαβαστούν μέσω στους ε, διάφορους αρμόδιους των θεσμικών οργάνων.